Τα θερμά μας συλληπιτήρια προς τα στις οικογένειες των θυμάτων των πρόσφατων θρησκευτικών ε, διώξεων και τρομοκρατικών επιθέσεων. Η γενοκτονία των χριστιανών δεν έχει πάψει. Μετά τη δολοφονία ενός ε, ιερέα στις Φιλιππίνες, χθες δέχτηκε επίθεση σε μια χριστιανική εκκλησία στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η οποία οδήγησε τουλάχιστον σε 10 θανάτους το κοινοβούλιο λέει φτάνει. Δεν μπορούμε να μένουμε αντρανείς και να βλέπουμε του ανθρώπους να διώκονται απλώς γιατί θέλουν να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Θέλουμε να συνεχίσει να ακούγεται η φωνή μας. και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν μπορούμε παρά να παραμένουμε σε επιφυλακή. Το δείχνουν οι επιθέσεις και οι σφαγές του Άιζη στο Αφγανιστάν και του Μπόκο Χαράμ στην Ιγυρία. Την Δευτέρα στην Καμπούλ είχαμε τρομοκρατικές επιθέσεις που προκάλεσαν 25 θανάτους, εκ των οποίων 11 παιδιά, 3 νεκροί ήταν και δημοσιογράφοι και ακτιβιστές ανθρωπιστικών οργανώσεων. Σε επίθεση στο τζαμί αγορά στην ε, Νιγηρία, η Μπόκο Χαράμ χθες ε, προκάλεσε τουλάχιστον 60 θανάτους αθώων. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια ένωση ολένα ισχυρότερη στο διεθνές προσκήνιο και έχουμε το στόχο να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία όσο περισσότερο μπορούμε προωθώντας την ειρήνη και τη σταθερότητα.